Uh, Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε νομίζω. Νομίζω ότι εδώ είναι όλες οι πολιτικές ομάδες. Θα χρησιμοποιήσουμε και την ψηφοφορία τις κάρτες μας για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εντάξει. Οπότε αν και εσείς όπως και εγώ έχετε ξεχάσει τη δικιά σας, φροντίστε να σας τη φέρει κάποιος όπως έκανα κι εγώ. Όταν χτυπάω εδώ το σφυρί μου, ακούγεται φοβερό τόρυβο εδώ, σε αυτό το έδρανο. Λέει ο πρόεδρο. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ για να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε σε μια πολύ σημαντική, πιστεύω, για μας συνεδρίαση, γιατί έχουμε να εξετάσουμε πολλές σημαντικές υποθέσεις. Όλοι σας έχετε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτές τους τελευταίους 12 μήνες, το οποίο αξιολογούμε όλους ιδιαίτερους και εκτιμούμε. Θα ψηφίσουμε και θα ακούσετε βέβαια και τους εισηγητές των, του συντάξεις μάλλον γνωμοδοτήσεων, που θα σας πούν δύο λόγια για αυτά που θα ψηφίσουμε αλλά μετά το καλωσόρισμα σε εσά, αλλά και σε όσους μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Εδώ έτσι κι δεν έχουμε πολύ χώρο στην αίθουσα, οπότε ίσως πολλοί να μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Θέλω να συμφωνήσετε πρώτα απ' όλα με κάποιες αλλαγές που έχουμε προβλέψει στην ημερήσια διάταξη. Η πρώτη αλλαγή έχει ως εξής. Για τις δημόσιες συμβάσεις έχουμε προβλέψει ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές να συνεδριάσουν και κλεισμένων των θυρών και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με αυτή την υπόθεση, μια που δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση προς το παρόν. Η πρόταση λοιπόν συγκεκριμένα λέει ότι θα συναντηθούν μετά την ψηφοφορία 12.30 με 1.30 αν βέβαια τελειώσει νωρίτερα η ψηφοφορία, μπορεί να αρχίσει νωρίτερα και αυτή η συνάντηση και κλεισμένο των ε, θυρών. Πιστεύω ότι είναι απολύτως λογικό. Δεύτερη αλλαγή. Βλέπω ότι είναι εδώ ο κύριος Φόξ. Κανονικά θα αρχίζαμε τη συζήτηση για την έκθεσή του όσον αφορά την αντίδρασή μας ε, στο έγγραφο της Επιτροπής για τα τυχερά παιχνίδια online το απόγευμα. Αλλά οι σκιώδες εισηγητές δεν θα μπορούν να είναι εδώ και εκείνος είπε ότι έχει κάποιες δυσκολίες. Γι' αυτό και επειδή πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, προτείνουμε να το αναβάλουμε για την επόμενη φορά που θα είναι όλοι εδώ. Δεν νομίζω ότι μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Ελπίζω να συμφωνείτε. Δεν ξέρω, ο κύριος Φόξ μήπως θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Καλώς. Τρίτον, τρίτη αλλαγή. Αύριο το απόγευμα Ακριβώς ε, πάλι επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι πάντα εδώ, αλλάζω την δικιά μου την ε, εισαγωγή όσον αφορά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων. Βέβαια ενημερώνεται και η Επιτροπή, ώστε να είναι εδώ η αρμόδια αξιωμετούχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, με τις αλλαγές αυτές ε, συμφωνείτε. Συνεπώς εγκρίνεται η διάταξη. Και πριν περάσουμε σε άλλα σημεία, θέλω να καλωσορίσω εδώ ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας, από ΤΑΛΚ, τον κύριο Μπόρισοφ, από τη Βουλγαρία. Χαιρετίστε, αν θέλετε, τους συναδέρφους. Καλώς ήρθατε. Παραδοσιακά σας καλωσορίζουμε με χειροκρότημα. Οπότε από εδώ και πέρα θα δουλεύετε μαζί μας προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Θα έχετε καλή εμπειρία σήμερα με την ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας. Στους φακέλους σας τώρα έχετε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2012. Αν δεν τεθεί κανένα ζήτημα, θεωρούνται εγκεκριμένα με τη λήξη της συνεδριάσεώς μας. Τι άλλο έχω να σας πω. Ότι έχουμε ένα νέο newsletter της Επιτροπής μας και υπάρχει και φωτογραφία όλων των μελών σε αυτό. Υπάρχουν αντίγραφα, μπορείτε να τα πάρετε. Και όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, αν θέλετε να ενημερώνεστε τακτικά, στείλτε μας ένα email και θα φροντίσουμε να σας το στέλνουμε. 2.000 άνθρωποι περίπου το παίρνουν με mail που ενδιαφέρονται στη δουλειά μας. Αυτό είναι πολύ καλό να το ξέρουμε. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι ο Ιρλανδός υπουργό θα έρθει αύριο, ο Ρίτσαρτ Μπρούτον, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την απασχόληση για την καινοτομία. Θα μας παρουσιάσει την Ιρλανδική Προεδρία. Α, όχι αύριο διορθώνει ο Πρόεδρος. Σήμερα, σήμερα, στις 3 θα είναι εδώ ο Υπουργός. Οπότε, σας παρακαλώ, Ακόμα και αν είσαστε κουρασμένοι από την ψηφοφορία του πρωινού, σας παρακαλώ να είσαστε εδώ στι 3 για να ακούσουμε τον κύριο Μπρούτον και να μπορέσουμε να τον ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε σχετικά με την Προεδρία. Περνάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο μας θέμα που έχουμε σήμερα, που είναι το πρόγραμμα τελωνίων. Ο κύριος Μπαλτασάρη είναι ο εισηγητής μας, σωστά. Είναι εδώ ο κύριος Μπαλτασάρη. Α, εδώ είσαστε, ναι, ναι. Κύριε Μπαλτασάρη, θέλετε να μας κάνετε κάποια εισαγωγή, όχι? Όχι, ωραία. Τότε να ψηφίσουμε ευθύ αμέσω. Για να πούμε τις λεπτομέρειες. Έχουμε ψηφίσει, θα θυμόσαστε, τα τελικά συμπεράσματα Συνεπώς, να αρχίζουμε. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία, έτσι. Όμως προηγουμένως να σας πω πού βρισκόμαστε. Οι τροπολογίες 10 και 13 του προπολογισμού έχουν καταπέσει. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 14 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην προπολογισμό 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προπολογισμό 16 και 17 καταπίπτουν. Προπολογισμοί 18 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Προπολογισμό 19. Καλύπτεται όμως. Οπότε περνάμε και ψηφίζουμε τώρα μαζί την 2, 3, 6 και 7 των προπολογισμών. Δεν έχετε αντίρρηση, έτσι. Ωραία. 2, 3, 6 και 7 προπολογισμών μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όμως την τελική πρόταση, παρακαλώ. Το τροποποιημένο κείμενο δηλαδή ψηφίζουμε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. 36 ψηφίζουν. Πέραστη τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 34 υπέρ, μία ψήφος κατά. Ευχαριστούμε κύριε Παλτασάρη, και συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στο πρώτο μεγάλο θέμα που έχουμε να ψηφίσουμε και που είναι η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Εδώ θα ζητήσω από την εισηγήτρια και αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, την κυρία Μπερναντέτ Βερνιό, να μας παρουσιάσει το θέμα της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλή σας μέρα όλοι. Θα ήθελα να αρχίσω με ευχαριστίες πρώτα απ' όλα προς όλους τους ε, σκιώδες εισηγητές και όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα. Είχαμε πραγματικά πολύ καλή συνεργασία για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα όλων των πλευρών. Επίσης, προκειμένου να προστατεύσουμε την απασχόληση μέσα στην εσωτερική αγορά. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα σε αυτήν την οικονομική και κοινωνική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, η κινητικότητα δεν είναι πολυτέλεια. Μερικές φορές είναι ανάγκη για πολλούς νέους, ιδιαίτερα από τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Συνεπώς, ο Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει την κινητικότητα αυτή να την διασφαλίσει και να την προστατεύσει περισσότερο. Ό,τι υπηρεσίε και αν είναι αυτές που προσφέρονται στους πολίτες. Ευχαριστώ επίσης τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και κυρίως την ομάδα μου εννοείται, αλλά και το ΕΛΚ, ΑΛΔΕ, ΓΚΟΕ, Πράσινη, CRFD, ε όλοι βοήθησαν. Μέχρι χτες αργά το βράδυ δουλεύαμε μαζί για να καταλήξουμε σε ένα κατάλογο ψηφοφορίας που να δείχνει ποιο είναι το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε όταν περάσουμε σε διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία, η οποία δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό για το θέμα και ε, παρόδο την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να μπορέσουμε να καταλήξουμε λοιπόν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε το όραμα του Κοινοβουλίου και έτσι να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλά. Δεν ξεχνά ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μαζί συνεργαστήκαμε πριν εμφανιστεί το κείμενο εκ παραλίλου, αλλά με τον κύριο Τίτσε και τους συνεργάτες του ε, συνεργαστήκαμε στενά για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κατάλογος ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε αργά, είναι αλήθεια. Στη σελίδα 88 και στην τροπολογία 706 πρέπει να σας πω ότι βάλαμε συν. Όσον αφορά την ομάδα μας θα πρέπει να είναι μείον. Να το ξαναπώ. Σελίδα 88. Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο 46, νέο. Άρθρο 58, παράγραφος 2, Τροπολογία 706 στη σελίδα 88. Σελίδα 88, 706 τροπολογία. Εντάξει, για μας πρέπει να λέει μείον εκεί, αντί για συν που έχει τώρα. Και μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία και σας ευχαριστώ όλους. Πρόεδρος, καλώς. Ωραία, θα αρχίσουμε. Εκτός αν κάποιος σκιώδης εισηγητής έχει να πει κάτι, αλλιώς μετά. Αρχίζουμε. Και όταν φτάσουμε στο σημείο που διευκρίνησε η Μπερναντέτ θα σας το πω, για να μην το ξεχάσετε. Πρόεδρε, δεν έχω τελειώσει όμως γιατί κάτι ξέχασα, κάτι πολύ σημαντικό. Διότι θέλω, υπογράμμισα μάλλον τη συνεργασία μας, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Την γραμματεία των ομάδων οι οποίοι, αν κατάλαβα καλά, δεν κοιμήθηκαν σήμερα τη νύχτα για να τα ετοιμάσουν όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα τον Σεμπαστιάν αλλά και όλη τη γραμματεία. Ξέρετε, είναι ακριβώ τα... οι κυφίνε, οι οποίοι, μάλλον συγγνώμη, είναι τα μερμηγκάκια τα οποία δουλεύουν σκληρά για να ε, κάνουν τη ε, δουλειά αυτή να γίνει πραγματικότητα. Υπέρ λοιπόν τη πρώτη, κατά, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρθρο 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 ε, περιβάλλοντος τώρα, ως προσθήκη. 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 10 περιβάλλοντος. Δεν ε, φαίνεται να δουλεύει η κάρτα μου. Τη βάζω, αλλά δεν ε, υπάρχει καμία αντίδραση από το μηχάνημα. Θα μεταφερθώ σε άλλο μηχάνημα. Ψηφίζεται υπέρ ή κατά. Υπέρ. Καλώς. Εγκρίνεται. 23 υπέρ και 13 κατά είναι το αποτέλεσμα. Ναι, και εγώ θα πήγαινα να καθίσω αλλού. Εγκρίνεται, είπαμε. Οπότε πάμε στη συμβαστική τροπολογία 30... 38. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 196 τροπολογία της κυρίας Ράπτη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 και 15 τώρα. Τις συγκήτρες υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνονται. Απασχόληση 18 καταπίπτει. 206 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Έληξε. 206. Της κυρίας Ρούλε. Για να επιταχύνουμε λίγο δεν βλέπω να έχετε ψηφίσει όλοι. Κύριε Μπρίντεγκα, τι συμβαίνει. Εκτό μικροφώνου, κύριε Μπρίντεγκα. Πέρα τη ψηφοφορία. Υπέρ ή κατά είσαστε. Υπέρ. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 19 κατά. Απορρίφθηκε, είπαμε. 21. Μακάρθιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 20. Απασχόλησης. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 205. Υπέρ. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και εδώ. Παρακαλώ, ψηφίζουμε για την τροπολογία Γούσταυσον 205. 38 ψήφισαν, η κυρία Μπρέντεκας είναι υπέρ, 19 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. έμβη 13. Και εδώ ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 13 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Γιατί είναι 19-19 το αποτέλεσμα. Δεν περνάει καμία. 209 τώρα της κυρίας Ρούλε. Πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 209. Πέρα στις ψηφοφορία. Κυρία Πρένικαρτ. Υπέρ. Ή, ή, μάλλον κατά. 23, 16. Εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει, λέει ο πρόεδρος. 17 καταπίπτει. Και τώρα πάμε στην τροπολογία. Καταπίπτουν οι επόμενες. Πάμε στην 18 της εισηγήτριας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 212 καταπίπτει. 19 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 της κυρίας Βακλάκη. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά νομίζω για την τροπολογία αυτή. Όχι. Α, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Απασχόλησης 22. Ηλεκτρονικά. Καλό θα ήταν αν φιλελεύθεροι δείχνανε τις προθέσεις τους πιο ξεκάθαρα, γιατί εγώ δεν βλέπω από τους φιλελεύθερους κανένα να ψηφίζει. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η κυρία Κέπαρτ και ο κύριο Σφαπ δείχνουν πώ ψηφίζουν. Οι φιλελεύθεροι δεν το δείχνουν. Ο κύριο Μπουζό είναι αυτό που το δείχνει. Καλώς. Να σηκώνετε πιο καλά το χέρι σα για να βλέπω. 214 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 215 και 11 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συνεπώς πάμε στην τροπολογία 291 της κυρίας Μακάρτιν. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 220. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 221. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 223 και 14 περιβάλλοντος υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περιβάλλοντος 15 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 228-229 περιβάλλοντος 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 227 καταπίπτει. 230 ως προσθήκη του κυρίου Αρίας. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Εγκρίνεται. Ε, Απασχόληση 23 τώρα, ως προστίκη. Πάλι ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε. Ο Κρίστιαν πώς ψηφίζει? Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Τροπολογία, είπαμε, απασχόληση 23 ως προστίκη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Έχω λάβει υπόψη μου και την κυρία Μπρέντεγκαρτ. 231 τώρα της κυρίας Μακλάρκιν. Υπέρ παρακαλώ, κατά, απορρίπτεται. 232. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 237. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 233. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 234. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 τώρα. 20. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 236. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεν την ψηφίζουμε. Οπότε πάμε στην περιβάλλοντος 17, 18, 19. Νομίζω ότι καταπίπτονται εφόσον έχει εγκριθεί 20 κάποια στιγμή. Σωστά. 20. Ναι. Επειδή εγκρίθηκε 20. Οπότε πάμε στην απασχόληση. Και η 239 καταπίπτει. Το 239. Υπέρ παρακαλώ, ως προσθήκη. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 240, 241, 242, 244, περιβάλλοντος 20, καταπίπτουν όλες αυτές, δεν τις ψηφίζουμε. και 21. 245 τώρα. Που είναι προφορική τροπολογία. Λεγκρίπ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 246 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 247 Να δω. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 247. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ και 15 κατά. 248. Μακλάρκιν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 250 και 249 καταπίπτουν και η περιβάλλοντος 21. 251 και 122 ψηφίζουμε τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 252 δεν ψηφίζουμε. 253 τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 255 καταπίπτουν και είμαστε τώρα στη 257 και στην ενβ 23 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. NV23 και 257. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, 20 κατά. Απασχόληση 28. Ψηφίζουμε τώρα υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απασχόληση 28 τροπολογία. 40 κάρτες υπάρχουν, αλλά 38 ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. 19-20. Τροπολογία 23 τώρα της εισηγήτριας. Υπέρ. 23 της εισηγήτριας. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά πάλι. 23 της εισηγήτριας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 18 κατά. Τώρα πάμε περιβάλλοντος 24, τροπολογία και 260 ως προσθήκη Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και επειδή εγκρίθηκε, πάμε στη σελίδα 18. 270. Μακλάκιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 285 καταπίπτει. 312, 278 τώρα και 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά. Όχι, ηλεκτρονικά μάλλον θα ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά. 256. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορία. απορριπτεται Απορρίπτεται. 20-20. Τροπολογία 27 της γύτρες υπέρ. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα η 280 και η NV29. Ως ε, προσθήκη πέρα, κατά, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 11. Εδώ κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Συμβαστική 11, πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Που είναι στην παράγραφο 5 της συμβαστικής. Υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα το ελέγξουμε αυτό. Ψηφίστε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 11. Πέρα τη φοφορίες, Εγκρίνεται από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, εντάξει. Το ΕΛΚ το αποφάσισε. Εγκρίθηκε. Οι επόμενες δύο σελίδες καταπίπτουν. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, οι τέσσερις μάλλον και έτσι φτάνουμε στην 313. Τι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 32 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 απασχόλησης, καταπίπτει. 314 Μακλάρκιν ως προσθήκη Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 315 ως προσθήκη Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. 317 τροπολογία. Ψηφίστε. Μόνο 37 ψηφίζουν από τους 40. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Με μία ψήφο διαφορά. Διορθώνει ο πρόεδρος. Μια που έχουμε και ένα μηχάνημα που δεν δουλεύει εδώ. 318 της κυρία Ζουρίλα. Ηλεκτρονικά. 318. που είναι ίδια με την περιβάλλοντος 35. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Συμβιβαστική 36 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 319 προσθήκη. Υπέρ. Κα... ηλεκτρονικά. 319 ως προσθήκη. Ψηφίστε. εγκρίνεται με 20 322 τώρα. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 33 της εισηγήτριας τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 33. Ψηφίστε. Πέρας της Απορρίπτεται. Συνεπώς. 35 προσθήκη της απασχόλησης, έτσι. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 323 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 39 περιβάλλοντος. Υπέρ. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα δούμε. Πολύ αργείται με την ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 25 ψηφί. υπέρ, 12 κατά. Τώρα έχουμε διάφορες ταυτόσιμες τροπολογίες, η NV38 για παράδειγμα και οι υπόλοιπε που είναι ίδιες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Γρήγορα με τις κάρτες σας παρακαλώ. Μην αργείτε τόσο. Γρήγορα. Πατάτε το κουμπί για να προχωράμε γρήγορα. Εγκρίνεται. Η 22 υπέρ 13 κατά. Άντε 23 μαζί με την, το μηχανό που δεν δουλεύει. Και τώρα υπάρχουν διάφορες που έχουν αποσυρθεί από τον κύριο Γούσταυσον. Και έτσι φτάνουμε στη συμβαστική 4. Συμβαστική 4. Κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το τμήμα 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2, προσψήφιση, υπέρ, κατά, εγκρίνεται επίσης. Όλες οι άλλες τώρα τροπολογίες καταπίπτουν και περνάμε τώρα στην τροπολογία 375 του εισηγητή. 375 του εισηγητή. Τη εισηγήτρια, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 375. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 18 υπέρ και 19 κατά. Τροπολογία 35 της εισηγήτριας υπέρ και εδώ νομίζω Τροπολογία 35 Είστε μαζί μου Τροπολογία 35 της εισηγήτριας υπέρ. Σηκώστε χέρια για να κάνουμε πιο γρήγορα. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Τροπολογία 43 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 373 και 3.74 ως προσθήκη υπέρ. Κυρία Φά, παρακαλώ, αποφασίστε. Ευχαριστώ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 376 της κυρίας Χέντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 377 και 378. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφώς απορρίπτεται. Τροπολογία 381 της κυρίας Ρούλε. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 379, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 380, υπέρ, κατά, αποχές, ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, θα... καλό θα ήταν να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται, νομίζω. Κλείνει ψηφοφορία. Σαφώς εγκρίνεται. Η 382 είναι συμβατή με αυτήν. Υπέρ λοιπόν η 382 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 383 της εισηγήτριας Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 383 έρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 19 κατά 18 υπέρ. 37 έχει αποσύρθει και περνάμε στην 384. Ποιος είναι υπέρ. 384 στην επόμενη σελίδα. Κατά. Όλοι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, εγκρίνεται. Εγκρίνεται σαφέστατα. Η 386 καταπίπτει. 388 τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 αποσύρεται. 389 της κυρίας Σάλντε Μεόζε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46 Επιτροπής Απασχόλησης καταπίπτει. Περνάμε στην 391. Τροπολογία 391. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 42 περιβάλλοντος καταπίπτεια ε. και η 390 επίσης, 47-48 επίσης, η 40 αποσύρεται. Περνάμε λοιπόν στην 395. 3.95 υπέρ κατά απορρίπτεται και μετά έχουμε μια σειρά από ίδιες τροπολογίες ξεκινώντας από την 3.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.93 από την κυρία Head υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.96 της κυρίας Ρούιλε υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται 397 υπέρ κατά και απορρίπτεται μαζί με την 50 της Επιτροπής Απασχόλησης τροπολογία 398 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 51 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά απο... απορρίπτεται 402 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 52 επιτρόπους απασχόλησης υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 401 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 403 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 404 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 400 καταπίπτει και η 399 είναι η επόμενη. Α, είναι συμβατή. Η 400, συγγνώμη, 400 είναι συμβατή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 400 εγκρίνεται, 399 είναι συμβατή. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 41 συμβατή από την εισηγήτρια υπέρ κατά εγκρίνεται. Μετά έχουμε την 53 απασχόλησης και άλλων υπέρ κατά απορρίπτεται. 407 και employment 54 υπέρ. Υπέρ λοιπόν 407 και 54 της Επιτρόπης Απασχόλησης να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19-19. Καταπίπτει. Απορρίφθηκε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε 37 κάρτες μέσα, δηλαδή περισσότερες κάρτες από όσους ψηφίζουν Δεν πειράζει. 42 λοιπόν όσος προστίκη από την εισηγήτρια υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 408 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 409 απορρίπτεται. 410 και NV43. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4-11 4-11 καταπίπτει και 4-12 4-12 καταπίπτει ή μάλλον όχι 4-12. τώρα να το ελέγξουμε ξεκινάει η ψηφοφορία για την 4-12. 40 κάρτες είναι τώρα μέσα αλλά 39 ψηφίζουν στην την κυρία πρεντεργκαστ πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται απορρίπτεται. 4-13 της κυρίας Μακλάρκεν Άρχεται η ψηφοφορία για την 4-13. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά στο ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Μπορείτε να είστε λίγο πιο γρήγοροι παρακαλώ. Κλείνει η ψηφοφορία. Τώρα έχουμε 41 εδώ. Εγκρίνεται. 4-14. Συμβατή. Υπέρ. Ε, πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τώρα έχουμε 40 που ψηφίζουν, 39 συν την κυρία Κλείνει η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 18 κατά. Τώρα σε μπλοκ 4-15 και λοιπές. Ας ελέγξουμε λοιπόν υπέρ, κατά, Έγκρινεται. Περνάμε τώρα στην έμπλα 55 υπέρ στη σελίδα 40. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 55. Κλείνει η ψηφοφορία. 18-18 και μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. κυρία Πρέντεργκας ψήφισε υπέρ, οπότε είναι 19, εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν η έμπλε 55. Περνάμε στην 4.17 και 4.18 ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Περνάμε στην 4.19, 4.20, 4.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 419, 420, 421 Περνάμε τώρα στην Επιτροπή Επασχόληση 56, ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 422 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 423, 425 υπέρ, κατά εγκρίνονται 424 καταπίπτει και 47 της Επιτροπής Περιβάλλοντος καταπίπτει επίσης και 43 είναι συμβατή με τις άλλες η 43 της Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. Κλείνει η ψηφοφορία. Η Απρέντεργας ήταν υπέρ. Εγκρίνεται με 20 υπέρ 19 κατά και μία αποχή. Αυτά λοιπόν για την τροπολογία 43, τροπολογία ε, ε, δετά υπέρ κατά απορρίπτεται, 58 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 428 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Κύριε Φόξ, σας ακούμε. Αυτή είναι η ομιλία του κύριου Κάμερον. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος ε, Πρωθυπουργός. Συμβαστική 39. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4.32 της κυρίας Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 433 της εισηγήτριας ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 434 της κυρίας Ρούιλε υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 435, 436 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 437 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 438 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 439 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 441 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 45 αποσύρεται, 442 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 60 απασχόληση υπέρ, α, καταπίπτει, συγγνώμη, 443 υπέρ, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.45 και MV48. Κύριε Μάντρες, παρακαλώ μην ενοχλείτε τον κύριο Σβάμπ, τον χρειάζομαι. 4.45 και MV48. Στην 46 πρέπει να ψηφίσουμε. Ας πάμε λοιπόν μία τροπολογία πίσω. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 46. 46 λοιπόν. Υπέρ. Θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 46. Ευχαριστούμε κυρία Πρέντερκα φροντίζουμε να έχουμε το μάτι μας πάνω σας. Ναι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 19 υπέρ 16 κατά. 46 εγκρίνεται. 4.45 λοιπόν και MV48. Και 4.45 λοιπόν. Είστε μαζί μου. 4.45. Χρειάζεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 20 16. 4-26. Τροπολογία 4-26. Συγγνώμη, εγκρίναμε την 445, οπότε καταπίπτει η 426. Σωστά. Περνάμε στην NV49 και τροπολογία 444 υπέρ, κατά, απορρίπτεται τροπολογίες 446 και επόμενες υπέρ κατά απορρίπτεται 449 υπέρ κατά εγκρίνεται 450 υπέρ κατά απορρίπτεται περνάμε στη συμβαστική 19 υπέρ κατά εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τροπολογία τη συμβιβαστική τροπολογία 24 υπέρ κατά εγκρίνεται περνάμε στην 460 και MV52 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 461 δεν τη θέτουμε σε ψηφοφορία 463 υπέρ κατά εγκρίνεται Περνάμε στην 50 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 464, 50 του εισηγητή. της εισηγήτριας, μόλις ψηφίσαμε την 50. 464 είναι συμβατή με την 50, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 53 περιβάλλοντος ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 465 αποσύρθηκε. 51 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 466 δεν θα ψηφιστεί. 52-53 της εισηγήτριας μαζί υπέρ κατά εγκρίνεται. 467 δεν θα ψηφίσουμε. Περνάμε στη συμβιβαστική 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Για τη συμβιβαστική. 33. Τμήμα 2 της συμβιβαστικής 33. Είναι σημαντικό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 33, τμήμα 2. Πέρας ψηφοφορίας Κυρία Πέντρεγκα ήταν κατά. Εγκρίνεται με 24 ενάντια 14. Και μία αποχή. Προχωράμε λοιπόν στην 495. Απευθείας στην 495. Δεν θα σα δίνω του αριθμού σελίδων γιατί διαφέρουν από αντίγραφο σε αντίγραφο. Τροπολογία 495 της κυρί... του κυρίου Μπουζόη. Ο κύριος Μπουζόη είναι υπέρ, σίγουρα. Δεν είναι σαφές, ας ανοίξουμε την ψηφοφορία γιατί είναι 495. Μπορώ να σας ζητήσω να ψηφίσετε πιο γρήγορα. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με 17 υπέρ, 22 κατά. 18, συγγνώμη, υπέρ. Περνάμε στην 496 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 504 του κ. Μπουζόη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογίες 05 και MV59 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 506 δεν θα ψηφιστεί. 507 υπέρ. Δεν είναι σαφές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 507. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ εγκρίνεται με 18 κατά. 508-509 δεν θα ψηφιστούν. 510 του κυρίου Μπουζόη. Υπέρ για την 510 κατά απορρίπτεται. 511 και MV60 υπέρ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για την 5, 11 και MV60. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 εναντί 18. 5-12 δεν θα την ψηφίσουμε. 5-13 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-14 και MV61. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 5-15 δεν ψηφίζουμε. Εμβι. 62. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5-16 δεν θα την ψηφίσουμε και περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 29 για τις ΜΕΣ υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς περνάμε λοιπόν κατευθείαν στην Εμβι. 64 διαγραφή υπέρ κατά Απορρίπτεται. 521. Δεν θα την ψηφίσουμε. 62 της εισηγήτριας. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ για την 62 της εισηγήτριας. Κατά. Εγκρίνεται. 528 έχει αποσυρθεί. 529 και 530 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 531 και 67. Κύριε Λίμπρο, ε, ψηφίστε για αυτή. Είναι στο τηλέφωνο, λέει. Νίκη ψηφοφορία, νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 19 υπέρ, 14 κατά. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στην 534 της κυρίας Ρούλε, υπέρ, κατά, υπέρ, συγγνώμη. Τις 534 θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας δυστυχώς απορρίφθηκε. 5.35 δεν θα ψηφίσουμε. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 32 με ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το τμήμα 1 της συμβαστικής 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 της συμβαστικής 32 Άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 2 της συμβαστικής 32. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται καθαρά. Παίρναμε στην 5-5-2, σωστά. 5-5-2. Τροπολογία διαγραφής υπέρ, κατά, ε, απορρίπτεται. 554 της κυρίας Ρούλε υπέρ. Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, φωνάζουν από κάτω. Περίμενα να μου κάνετε σήμα 5-5-4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5-5-5 Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική 20. Συμβιβαστική 20. Είμαστε στη συμβιβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 568 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 568 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνάμε στην 569 ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 570 καταπίπτει. Περνάμε στην 572. Τροπολογία 572. Να δω χέρια. Υπέρ της 572. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 22. Υπέρ κατά εγκρίνεται περνάμε στη συμβεστική 23 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 580 υπέρ κατά εγκρίνεται 564 υπέρ κατά εγκρίνεται 581 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 582 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 583 δεν θα την ψηφίσουμε. 584 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 585 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 περιβάλλοντος και λοιπές όμοιες ε, τροπολογίες υπέρ κατά επίσης απορρίπτονται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 590 της κυρίας Τούρνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 της ε, Επιτροπής Αποσχόλησης υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 591 ως προσθήκη. Υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ως προσθήκη. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 17 περί 22 κατά 594 και 78 υπέρ κατά εγκρίνεται. 593 την προσπερνάμε. Τώρα είμαστε στην 595. Υπέρ και κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν πάμε στην 621 Τροπολογίε διαγραφή. Αυτέ λοιπόν από τι 6.21 υπέρ, κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην συνδυαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Κατά. εγκρίνεται. Τροπολογία 6.22 του εισηγητή, υπέρ, κατά απορρίπτεται. Η 75 έχει αποσυρθεί. 6.43 και 6.76. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.42 της κυρίας Μακλάρκιν, υπέρ, κατά, απορρίπτεται και αυτή. Τώρα, συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν. Ε, τροπολογία σε μπλοκ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπέρ. Θα πρέπει να ανοίξουμε την ψηφοφορία. Ένβη 86 έως 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 78, 79, 84... 6.43 καταπίπτει. 6.53 καταπίπτει, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 14 τώρα. Συμφωνούμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 664 της κυρίας Τούρουνεν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 665 Θέλετε να τις κάνουμε σε πλό, κύριε Τούρνεν. Νομίζω πως κάποιες ομάδες θέλουν να ψηφίσουν, γι' αυτό θα τις πάμε μία-μία. 6-6-5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-6-6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 668 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 670 και NV96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 669 την προσπερνάμε 671 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 673 Νομίζω πως πάλι θέλουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 6.73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6.72 ως προσθήκη. Ψηφίζουν οι φιλελεύθεροι. ηλεκτρονική ψηφοφορία. 6.72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφους και 18 κατά. Ήθελα να δω πώς ψήφισε η κυρία Πρένταρκας. Λοιπόν, 6.74 της κυρίας Ρούλε. Υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. Λοιπόν, να σε ελέγξουμε. Α, πέρας πληροφορίας, 24 υπέρ, 16 κατά. 6,75. Κυρία Τούρουνεν, υπέρ. Πρέπει να κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. 6.75 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Είναι 20 και 20. Καταπίπτει. 83 της συγγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6.77 της κυρίας Ρούλε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 6.78 κυρία Βάσκεμπα και άλλοι. Είστε υπέρ ή αλλάξατε τη γνώμη. 678. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84 της εισηγήτριας. 679 της κυρίας Ράπτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 85 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 682 της κυρίας Βάισκεδα. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 680 της κυρίας Ρούλε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται κι αυτή. 681 σε ένα λοβά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 684 υπέρ να κοιτάξουμε ηλεκτρονικά την 684. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψηφικάτα απορρίπτεται. 685 προσθήκη της κυρίας Βάις Κέρπερ. Ψηφίζουν οι φιλελεύθεροι. Υπέρ. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 ψήφι υπέρ, 16 κατά. 686 της κυρίας Ρούλε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 6,90 και employment 80 υπέρ. Θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Και οι δύο εγκρίνονται. 689. Προηγούμενες καταπίπτουν ως προσθήκη. 689. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Employment 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε ψηφοφορία σε μπλοκ για τις έξι τροπολογίες της κυρίας Ρούλη από, τις, από την 699-696 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται όλες. 693 Άριας υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 700 και 701 της κυρίας Πετικάινεν. Σας καλωσορίζω. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Πάνω στην ώρα ήρθατε. 703 της κυρίας Πρέντεγκαστ. Όχι, οι προηγούμενε καταπίπτουν, λέει ο πρόεδρο. Είμαστε στην 704. Η 703 εγκρίνεται. 706. Μισό λεπτό να κοιτάξουμε. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, κοιτούσαμε να δούμε που βρισκόμαστε. Ποιες τροπολογίες καταπίπτουν. Λοιπόν, το κοιτάξαμε γιατί δεν ήμασταν σίγουροι τι γίνεται με την 704. Μάλιστα. Προχωράμε στην 706. όπου άλλαξε η άποψη της εισηγήτρες. Λοιπόν, 706 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 707, 708, 709 δεν θα ψηφιστούν. Γι' αυτό προχωράμε στην 712 και 713. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα στην, για την τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7-14. Είναι συμβατή με. Αυτό υπέρ. Ας κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για την 7-14. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 υπέρ, 18 κατά. Η 7-15 είναι επίσης συμβατή. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 716 καταπίπτει. Διότι 7-12 εγκρίθηκε. Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε. 716. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 717, 718. Δεν θα τις ψηφίσουμε. 719 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 720. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 7.20. Δεν μπορούμε να το δούμε αλλιώς. 19 υπέρ 20 κατά, μία ψήφος απορρίπτεται. Καλά κάναμε και το κοιτάξαμε. 721 υπέρ κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 722. Κύριε Γκάλπελτς, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 720 έχει αποσυρθεί. Περιβάλλον 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Employment 1 γιατί NV6 καταπίπτει employment 1. Ας κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Employment 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 93. Συμβατή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. NV2 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 90 και 96 καταπίπτουν employment 2 υπέρ, Νομίζω πως πρέπει και εδώ να κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, 19-19, employment 3. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Σχεδόν στην αρχή γυρίσαμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1 στο αιτιολογική σκέψη 4. Είμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ. Και είναι κατά. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 108 της κυρίας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα στην βαστική τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117. Αιτιολογική σκέψη 80. Διαγραφή υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 119. Κυρία Τούρουνεν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Employment 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Employment 8 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 121, κυρία Ρούλε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 121 της κυρίας Ρούλε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 122 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 126 της κυρίας Βάιλερ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της εισηγητρίας, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131 τώρα. Οι προηγούμενες καταπίπτουν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Χέρια παρακαλώ. Ναι, εσείς και ο κύριος Φαμπ διαφωνείτε. Κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και 152 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 23, 160 τροπολογία υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, ας κοιτάξουμε ηλεκτρονικά, 159, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 171 Ένα, του κύριου Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 172. Κυρία Ρούλε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174. Κυρία Ρούλε. Υπέρ. Ας κοιτάξουμε τις τροπολογίες της κυρίας Ρούλε οριστικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Μία ψήφος παραπάνω κατά. Οριστική ψηφοφορία κυρίες και κύριοι. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Θέλει κάποιος άλλος να ψηφίσει. Κυρία Πρέντερ, είστε υπέρ. Όλοι έχετε τις κάρτες σας. Κάποιος ψηφίζει τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι, 33 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. κυρία Ρούλε, νομίζω πως έχει το δικαίωμα να πει μερικά λόγια. Όχι, κυρία Βερνιό, συγγνώμη. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Μετά την ψηφοφορία διαπιστώνουμε ότι πολλές ε, τροπολογίες ψηφίστηκαν με πολύ μικρή διαφορά. Νομίζω όμως ότι έχουμε καταλήξει σε μια πλειοψηφία μεταξύ μας και θα αρχίσουν έτσι οι διαπραγματεύσεις πια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την δουλειά προκειμένου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση από πάνω ώστε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σχέδιο για τους πολίτες από τους επαγγελματίες. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω όλους σας. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μιλήσει, όχι συγγητές. Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα. Προτείνω να κάνουμε ένα λιγό λεπτό διάλειμμα ανάμεσα στις ψηφοφορίες. Τεντωθείτε και μετά επιστρέφουμε με την έκθεση του κυρίου Σφάμπ. Μπορείτε να σηκωθείτε λίγο Uh, so, um, Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τη συγκέντρωση και την προσοχή που έχετε δείξει στη μεγάλη ψηφοφορία για την αμοιβή αναγνώριση. Έχουμε τρεις άλλους φακέλους να ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να με βοηθήσετε και να συνεχίσετε να είστε προσεκτικοί. Κύριε Σφάμπ, θέλω να μου δώσετε το σήμα σας να ευχαριστήσω τους ε, συντονιστές και αν έχω μία ένδειξη για τις θέσεις σας μπορώ να κάνω την ψηφοφορία πιο γρήγορη, να ελαχιστοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην έκθεση του κυρίου Σβάμπ για συστάσεις για διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Κύριε Σφάμπ, θέλετε να πείτε μερικά πράγματα. Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της ομάδας μου το βραβείο που λάβατε, στο, το CBE δηλαδή, στο Ενωμένο Βασίλειο. Και ο David Κάμερον είπε ότι η Βρετανία θα παραμείνει στην ενιαία αγορά, οπότε νομίζω πως αυτό βοήθησε, θα μας πάει πιο μπροστά. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία. Ε, με χαροποίησε πάρα πολύ το ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ενίες θέσεις για όλα σχεδόν τα θέματα. Ενσωματώσαμε και τις συμβολές των άλλων επιτροπών και ως Επιτροπή είμαστε μία από τις ελάχιστες η οποία τώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει δώσει, δίνει τώρα μία γνωμοδότηση η οποία μπορεί να υποστηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες και το βρίσκω πολύ θετικό και ελπίζω να μπορέσουμε μαζί να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε στο να γίνει η ενή αγορά ένα σημαντικό στατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο επόμενο ερώτημα είναι ποια νομική βάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση. Εδώ έγινε συνέντε... συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω εδώ τις ειδικέ επιστημονικές ομάδες του Κοινοβουλίου που μας έκαναν τις μελέτες. Πρέπει να βρούμε επιχειρήματα με τα οποία να μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για τα επιχειρήματά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας όλους. Well, thank you very much, Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τις ευχές σας και καθώς ε, και για την εργασία σας σε αυτόν τον φάκελο. Συμφωνώ μαζί σας, είναι εξαιρετικά σημαντική η δουλειά που κάνουμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Αρχίζουμε με συμβαστική τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ένα του κυρίου Ντεγιόγκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία, όπως βλέπετε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δύο, της κυρία Κοράτσα Μπίλτ, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Όχι, είναι, υπάρχει μια προφορική τροπολογία, λέει ο πρόεδρο. Συμβιβαστική τροπολογία 1, χωρίς τις προφορικέ τροπολογίε. Συμβιβαστική τροπολογία 1, με τις προφορικές τροπολογίες υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συμβιβαστική ένα με τις προφορικές μαζί. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε. Τώρα λοιπόν, συμβιβαστική τροπολογία 1 χωρίς τις προφορικές. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα συμβιβαστική 1 χωρίς τις προφορικές. Προχωρούμε τώρα στην τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Employment 3 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική τροπολογία 26. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21. Καταπίπτει 21. Ψηφίζουμε λοιπόν τις προφορικές τροπολογίες. Την προφορική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Employment 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 23 έχει αποσυρθεί, 24 του κυρίου Ντεγιόν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 25. 5, λέει ο πρόεδρο. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβιβαστική τροπολογία 24. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και συμβιβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επιτροπή Ρέτζι 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 23 εγκρίθηκε, άρα η 133 καταπίπτει. Τροπολογία 36, κύριο Κοφεράτη, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 37 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, εγκρίνεται. 39. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 40. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 40 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κυρία Σολτεμόζε, ήρθατε στην ώρα. 41 ως προσθήκη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 48. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται κι αυτή. Η 50 καταπίπτει, η 51 τώρα. Υπέρ, κατά, Δεν είναι ξεκάθαρο. 51. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 19 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Να ελέγξουμε για την 61 παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. 61. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. διαφορά. 19-18. Συμβιβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. συμβιβαστικη 17 υπερ κατα εγκρινεται Εγκρίνεται. Τροπολογία 135 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Να δω. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα του κυρίου Σβάπ και Κοφεράτη επί της 77 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. 78. Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79. 79. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε 81 Ογδόντα ένα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 20-16. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται η Α, όχι, εγκρίνεται, σαφώς. Εγκρίνεται λοιπόν σαφώς. 83 είναι η επόμενη. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά εγκρίνεται 1.45 κρύο που πάει και υπέρ κατά εγκρίνεται και 1.46 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά εγκρίνεται και τροπολογία 149 που δεν ε, μπει στο συμβεβασμό υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 1.54 υπέρ 1.54 1.54 υπέρ κατά εγκρίνεται περνάμε στην 1.56 υπέρ κατά κατά εγκρίνεται 1.57 καταπίπτει 86 υπέρ κατά εγκρίνεται 88 ε, το κύριο Κοφεράτη υπέρ κατά εγκρίνεται 89 υπέρ κατά εγκρίνεται 90 υπέρ θα χρειάζεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά 18 υπέρ 19 κατά. Απορρίπτεται συνεπώς. Περνάμε τώρα στην συμβεβαστική 20. Στα παρατήματα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ. Πώς ψηφίζουν οι φιλελεύθεροι για αυτήν. Να ανοίξουμε την ψηφοφορία. Δεν είναι καθόλου σαφές. είμαστε στην, 80, στην 96 συγγνώμη, τροπολογία αυτή τη στιγμή. Τροπολογία 96. Κλείσατε την ψηφοφορία πολύ γρήγορα. Την επαναλαμβάνουμε από την αρχή. 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Είστε πολύ αργοί αυτή τη στιγμή. Κλείνει η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Εγκρίνεται σαφώ. 97 έχει αποσυρθεί. Προφορική για την παράγραφο 4 του κ. Σβάμπ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 98 του κ. Ντεγιόγκ υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ κατά εγκρίνεται 101 υπέρ κατά απορρίπτεται 1, 01, 103, 02, 03, 104, 105 δεν θα τις ψηφίσουμε Περνάμε στην 106 προφορική τροπολογία περ. Κατά. Εγκρίνεται. 107 προφορική τροπολογία του παραρτήματο 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107 τη κυρία Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108 του κυρίου Κοφεράτη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109 τεχνική τροπολογία 110 του κ. Ντεγιόγκ υπέρ κατά απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά απορρίπτεται. 112 της κυρίας Κορατσαμπίλτ υπέρ κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβεβαστική 36 υπέρ κατά εγκρίνεται. 114, διαγραφή της κυρίας Μακλάρκιν, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 115 ε, του κ. Κοφεράτη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 21 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 119 διαγραφή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 120 του κ. Ντεγιόγκ υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, εγκρίνεται 121 υπέρ κατά εγκρίνεται 122 υπέρ κατά εγκρίνεται 123 έχει αποσυρθεί 159 είναι συμβιβαστική 124 όχι 125 επίσης καταπίπτει νομίζω 126. Πρέπει να ψηφίσουμε την 126 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβεστική 37 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τέλος, 128 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία για το συνολικό ψήφισμα πέρας ψηφοφορίας 33 υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σφάμπ Να, ένα χειροκρότημα σας αξίζει. Κύριε Σφάμπ, θέλατε να πείτε κάτι για το ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του σημαντικού ψηφίσματος και πώς θα συνεχίσουμε με αυτή την ίδια πρωτοβουλία. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, θα έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Η διακυβέρνηση της νέας αγοράς και η έκθεση αυτή είναι συστατικό στοιχείο μιας κοινοβουλευτικής απάντησης στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ως απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει και τον ίδιο τίτλο. Οι συντονιστές όμως αποφάσισταν, κύριε Πρόεδρε, να συμπεριληφθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενίας Αγοράς για ολοκλήρωση, τη γνωμοδότηση για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς. Γι' αυτό το επόμενο βήμα θα έχει ως εξή. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο ως Επιτροπή να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μια κανονική γνωμοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις ε, προτάσεις μας για την βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς και να συνεργαστούμε δημιουργικά έτσι ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική πρόταση. Very briefly. Ε, εν συντομία ήθελα να σας συγχαρώ. Θα γίνετε πραγματικός ε, Βρετανός. Ε, όλοι έχουν λάβει τιμές, σήματα τιμής. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω για τον Κάμερον για σήμερα το πρωί και για που σχετίζεται με αυτή την έκθεση ότι ο Κάμερον υποστήριξε την ύπαρξη ε, ενό τμήματο για την αγορά, για την ενιαία αγορά. Είπε ότι η ενιαία αγορά είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει σύνοδο κορυφή των Υπουργών Ενιαία Αγορά. Έχουμε για τι μεταφορέ και για άλλου τομεί. Δηλαδή, η Επιτροπή μα θα έπρεπε να εστιαστεί περισσότερο στην ενιαία αγορά και στην πρόθεση τη. Περισσότερο από ό,τι ακόμη και από ό,τι και σήμερα. That's Πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα που λέτε. Πολύ χαίρομαι που το ανέφερε ο κύριος Κάμερον στην ομιλία του. Κυρία Καπάτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για το νέο τίτλο τιμής που αποκτήσατε. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε μία εξέχουσα προσωπικότητα ανάμεσά μας. Να συγχαρώ επίσης και την, το κύριο Σφάπ και την έκθεση την οποία ψηφίσαμε. Χαίρομαι πολύ που η ιδέα που εισήγαγε η ομάδα των ε, Σοσιαλδημοκρατών στην ε, συνάντηση των συντονιστών υιοθετήθηκε ως συστατικό στοιχείο στην έκθεση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και φαίνεται πως τώρα έχει ολοκληρωθεί το θέμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό διότι θα ήταν ε, μη αποδεκτό από εμάς οι, οικονομίες, οι επιτροπές ΕΚΟΝ και έμπλη να μην είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Δεν έχει μόνο όμως να κάνει έκθεση με την ε, οικονομική διάσταση, αλλά και με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιχειρήσεις. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και να θέσουμε τους πολίτες στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι κάτι που για μας τους σοσιαλδημοκράτες είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ακριβώς ε, για αυτό το λόγο, επειδή ήταν μέρος της έκθεσης, μπορούσαμε να το υπερψηφίσουμε και ελπίζω η δουλειά που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μια πνοή ανέμου στην βελτίωση της διακυβέρνησης. Και ελπίζω να συνεχίσουμε ως σοσιαλδημοκράτες να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Good. I think we're... Ωραία, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα της έκθεσης του κυρίου Μπερτ για την ευρωπαϊκή αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον Γιάννη Άντερσον. Πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ ήρθατε να δείτε τι δουλειά κάνουν οι διαδοχοί σας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μας επισκέπτεστε. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε και περνάμε σε μια σημαντική γνωμοδότηση όσον αφορά την ε, προστασία δεδομένων. Είμαστε η πρώτη επιτροπή που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει δηλαδή το βαθμό ενδιαφέροντος Πόσο πολύ δηλαδή ενδιαφέρεται η Επιτροπή μας για αυτά τα θέματα. Η κυρία Κόμη ίσως θέλει να πει δύο λόγια πριν την ψηφοφορία. Ε, κύριε Σφάμπ και εσείς, γι' αυτό, α, όχι για το προηγούμενο, γι' αυτό. Ωραία. Η συγκίτρια όμως πρώτα, παρακαλώ, να πει δύο λόγια και μετά να ψηφίσουμε. Η Λαρακόμη έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, τους κοιόδης διότι αληθεύει αυτή η γνωμοδότηση δίνει πολύ σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ε, προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ε, έχουμε προβλέψει και την ψηφοφορία κιόλα, διότι το σχέδιο έκθεση στη Λίμπε παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες. Συνεπώς ήμασταν πολύ γρήγοροι και αυτό περιλαμβάνει διάφορα υπέρ και κατά, αλλά πιστεύω η δουλειά που κάναμε θα είναι ωφέλιμη. Θα συνεργαστούμε στενά και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και τις λοιπές ε, επιτροπές και στους τριμερείς διαλόγους, διότι αυτό αφορά κυρίως την εναρμόνιση ενός συστήματος και αυτό το έχουμε αναδείξει και το έχουμε επισημάνει σε, πολλές, σε πολλές έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τις Σκιώδης προνόμιο ήταν για μένα να είμαι και εγώ σκιώδης ε, εισηγητής. Κύριε Σφαμπ, τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για τη δουλειά της. Όμως, ε, για να καταλάβουμε καλά την θεσμική κατάσταση, Πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την εισηγήτρια να ετοιμάσει την ανάλυση της για μια έκθεση η στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακόμα. Οπότε εδώ τίθεται θέμα συνεργασία με την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να καταλήγει σε φαρσοκομωδία αυτή η υπόθεση. Οπότε από πλευρά μα μπορούμε να πούμε ότι με την έκθεσή μα θέλουμε να συνεισφέρουμε σημαντικά, αλλά τελικά δουλεύουμε μέσα σε κενό. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Λίμπε. Νομίζω ότι στη διάσκεψη των Πρόεδρων πρέπει να το θέσετε, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, καλώς. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ναι, σε έναν βαθμό. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να επηρεάσουμε. Γι' αυτό, έτσι κι αυτό πρέπει να κάνει μια καλή γνωμοδότηση. Κυρία Σαντομόσα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Αλλά πρέπει να πω πως σήμερα όταν θα φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Εξαρτάται από το πώς θα έχει προχωρήσει η ψηφοφορία μέχρι τότε. Σίγουρα είχαμε καλές συζητήσεις, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα υπερψηφίσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία κλειδί για μας τα θέματα για την παραβίαση, το πόρο του δεδομένου και άλλα. Οπότε εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία, ποια θα είναι η τελική μας θέση, στην τελική ψηφοφορία δηλαδή. Οι συζητήσεις ήταν σίγουρα πολύ καλές και θα προσπαθήσουμε και εμείς να επηρεάσουμε την ΛΥΜΠΕ για τις παρετέρω εργασίες της. Πρόεδρος. Ωραία, πριν την τελική ψηφοφορία, ωραία, θα σας δώσω τη δυνατότητα να το συστήσετε μεταξύ σας. Το καταλαβαίνω. Ωραία, ψηφίζουμε. Εκτός αν θέλει κανένα άλλο το λόγο, όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. Τροπολογία 147. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να βεβαιωθούμε, να δούμε και ποιοι είναι εδώ ποιοι δεν είναι, πώς ψηφίζουν οι ε, διάφοροι. Ηλεκτρονικά λοιπόν, 147 ψηφίστε. «37 κάρτες υπάρχουν, 31 ε, ψηφίζουν». Εγκρίνεται πάντως 21 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. 148 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 149 ως προσθήκη. Υπέρ. Οι φιλελεύθεροι να μου δείχνουν τι ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν. Κατά. Εγκρίνεται. 150 κατά πίπτη. 151. Σασκόφσκι. Υπέρ. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 153. Τρασκόφσκι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 155. Όχι, 154 λέει πάλι ο πρόεδρο υπέρ. Για να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. 155. Στήλερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Ας ελέγξουμε. 157. Ψηφίζεται διαφορετικά, με διαφορετικούς συνασπισμούς σε κάθε τροπολογία, οπότε μου είναι δύσκολο να προβλέψω τα αποτελέσματα. Εδώ έχουμε 16-17, οπότε απορρίπτεται. Τροπολογία 30 της εισηγήτριας τώρα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 158, Λεκεγκάρτ. Υπέρ. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε. 158. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται. 19 υπέρ 16 κατά. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 32 έχει αποσυρθεί. 165 λέει και γάρτη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 169 και 170 που είναι ίδιες υπέρ. Θα αλλάξουμε ηλεκτρονικά. 169 και 170. Ψηφίστε. Και πιο γρήγορα παρακαλώ. Μην περιμένουμε τόση ώρα. 18 υπέρ, 17 κατά εγκρίνονται. 171 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 171. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρες της ψηφοφορίας. 18-16 εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 176 και 178 έχουν αποσυρθεί, 177 ως προσθήκη του κύριου Λούκεγάρτ. Υπέρ παρακαλώ. Δεν είναι ξεκάθαρο. 177. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. 19-16. Εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά δεν καταλαβαίνω 180 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε πέρας υποφορίες, εγκρίνεται 19 μάλλον 16 ναι, 19-16. 179 ναι, και 34 καταπίπτουν, 181 και 35 έχουν προσθέσει, 183 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίστε. 182. Πέρες υποφορια εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 185. Στάιλερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αλλά μάλλον να το ελέγξουμε γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 19 κατά. Απορρίπτεται. Δεκαπέντε υπέρ, 19 κατά. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187 κατά πίπτη, 188 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 18-15. Εγκρίνεται. 189. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε με 189. Τσίμα τσίμα μου φαίνεται το αποτέλεσμα. Ψηφίστε. 189. Απορρίπτεται. Αν είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σας, θα πάμε πιο γρήγορα. 191, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 190 καταπίπτει. Α, όχι. 190. Ως προσθήκη την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 194. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά. Για να ελέγξουμε. Να πούνε και δικιά μου τροπολογία, να μην έχουμε αμφιβολίες. Μην νομίζετε ότι είμαι προκατηλημένος δηλαδή γι' αυτό. Εγκρίνεται από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ. 197. Λεκεμπερ. Κάρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 200. πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία Σαλβίνη. Τώρα, τροπολογία 36, 201, 202 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 203 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 204. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 205. γάρτα, αλλά κατά τμήματα ψηφοφορία έχει ζητήσει το ΕΛΚ. Συνεπώ, ψηφίζουμε το πρώτο μέρο. Υπέρ, παρακαλώ, του πρώτου τμήματο. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καταπίπτουν 207, 37, 206 είχε αποσυρθεί, 208 καταπίπτει, 209 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 210. Υπέρ. Θα ελέγξουμε. 210 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα της φοφορίας, Εγκρίνεται. 211 καταπίπτει, συνεπώς 212. Όχι, δεν την ψηφίζουμε. Ε, όχι, την ψηφίζουμε. 212. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 213. Έγκστρομ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 214. Σάντερ Μόζο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 224. Α, ναι, tips. Κύριε Κοράτσα Θέλετε χωριστά να ψηφιστεί 220 και όχι δεν θεωρείτε ότι καλύπτεται από τη συμβιβαστική και τη θέλετε ως προστίκη. Συμφωνείτε όλοι να την ψηφίσουμε χωριστά. Ωραία, 220 λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ευχαριστώ κυρία Κορατσαμπίλτ. 224, λέω και καρτή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 225 ως προστίκη της κυρία Στάιλερ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 229 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 230 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 231 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά εγκρίνεται. 234 υπέρ πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για τη 234 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 16 κατά, 18 υπέρ, μία αποχή. Εγκρίνεται. 235 τότε. Υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε για τη 235. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 20 υπέρ 14 κατά. Εγκρίνεται. 236 προσθήκη στην 235 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 237 υπέρ πρέπει να ελέγξουμε. Γιατί το ΕΛΚ φαίνεται να έχει διαφορετική, να είναι διχασμένο. 237. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίστε. ...30 υπέρ, 5 κατά. 238 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 240 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αλλά ίσως καλύτερα να το ελέγξουμε και αυτό, γιατί πολύ τσιματσίμα μου φαίνεται. Ψηφίστε 18 υπέρ, 16 κατά. Πραγματικά πολύ τσιματσίμα, καλά έκανα και το ήλεγξα. Και έτσι η δικιά μου καταπίπτει. Ε, και η 239. 241 ως προσθήκη λοιπόν της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 245 καταπίπτει. 246 Λέγκαρτ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 247 Τρασκόφσκι υπέρ. Θα το ελέγξουμε. 247. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 18 υπέρ και 16 κατά. Και μία αποχή. 249 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 248 ως προσθήκη της Κεντεβερνιό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 250 υπέρ. Θα ελέγξουμε. 250 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίες. Απορρίπτεται. 18 κατά. Ε, λυπάμαι που παίρνω το λόγο τώρα για το 17, όμως θυμάμαι ότι στην τελευταία ψηφοφορία, στην άλλη αίθουσα, εσείς κυρία συνάδελφοι, δεν είχατε την κάρτα και αρνηθήκατε λοιπόν την ψηφοφορία. Σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα με την κυρία Πρέντεγκαστ, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω αύριο στην ψηφοφορία να γίνουν αποδεκτά μόνο αποτελέσματα που θα έχουν ε, γίνει με ηλεκτρονική κάρτα, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Κύριε συνάδελφε Σφαμπ, η κυρία Πρέντεκαστ είχε την κάρτα της, η κάρτα δεν λειτουργούσε όμως. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε λοιπόν για αυτό το πράγμα. Δεν κατηγόρησε, λέει ο κύριο Σφαμπ. Απλά να παρακαλέσω αύριο στην ψηφοφορία να διαβεβαιώσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί. Well, Mrs. Πρόεδρος, η κυρία Πρέντεκαστ θα προσπαθήσει να βρει μια άλλη. Μου την έδειξε. Όντω την έχει. Δεν βάζει την κάρτα επιβίβαση αντί για την σωστή. Απλώς δεν δουλεύει η κάρτα της, το έχω ελέγξει και εγώ. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε μέχρι αύριο. Αλλά και εσείς φροντίστε να έχετε όλα σας τα μέλη εδώ. Μερικές φορές είναι πολύ τσιματσίμα τα αποτελέσματα επειδή δεν είναι όλοι εδώ. Αν όλοι κάνουμε μια προσπάθεια, ίσως να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, πού ήμασταν, 251. 251. Ψήφι. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. 251. Αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και εδώ. Για να είμαι σίγουρος ότι μετράω όλες τις ψήφους. 21 ψήφοι υπέρ, 14 κατά με το μηχάνημα που δεν δουλεύει. 252, Στάιλερ. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Για τη 252. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ 20 κατά. 39 έχει αποσυρθεί. 253 και 254. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. 40. Κόμι. Υπέρ παρακαλώ. Για να ξαναδώ τα υπέρ. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 15 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. 255 πίπτη ή όχι. Όχι. Α, ναι. Η 40 πίπτη. 255 τώρα. Υπέρ. Κατά. θα πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό. Ηλεκτρονικά, έτσι. Πέρα τη φοφοριες εγκρινεται Εγκρίνεται. 19-16. 41 της εισηγητρίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 256 και γάρτη. υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 257 Τρασκόφσκι. Ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. το αποτέλεσμα απορρίπτεται. 42 έχει αποσυρθεί. 258. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43. Τη συζήτηση υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 259. Τρασκόφσκι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 261. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 260. Ε, ως προσθήκη. Υπέρ της προσθήκης. Κατά. Εγκρίνεται. 44 ακόμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 280. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 281. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 284 καταπίπτει είπαμε. Α, τη 41 μόλις την ψηφίσαμε. Α, όχι, τώρα ψηφίζουμε λέει τη 49 της εισηγήτριας, υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις προφορίες. 17-17 το αποτέλεσμα απορρίπτεται. Τώρα 285 του κ. Τεταφυλίδη. Υπέρ. Θα ελέγξουμε. 285. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. 286. Υπέρ. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για τη 286. Πέρας της υποφοριας εγκρινεται Εγκρίνεται. 20-16. 287. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 50 έχει αποσυρθεί. 288 Τρασκόφσκι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 289. Α. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για τη συμβαστική τροπολογία 9. Ψηφίστε παρακαλώ. 20 υπέρ, 15 κατά μια εποχή. 320 τώρα. 320 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 και 322 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 324 υπέρ, Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 324. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. 323 κατά πίπτη, 325 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 328 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 326 και 55 καταπίπτουν συνεπώς. Ή την προσθήκη. Όχι. Και 327 καταπίπτει. Συνεπώς, 329 και 330 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνονται. 331 και 332 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 56 της κυρίας Κόμη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57 έχει αποσυρθεί, 333 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 338 υπέρ θα ελέγξουμε εδώ. 338 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 20 υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. 337 καταπίπτει, Συνεπώ 339 τώρα υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 340 καταπίπτει, 341 λοιπόν υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 346 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ, να ελέγξουμε καλύτερα εδώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. 347. Πέρας στις ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16-18. Είχε αποσυρθεί 60, 61 και 348 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 350 έχει αποσυρθεί. 351 και 352 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε καλύτερα. Προτιμάω να που είναι και συμβαστική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τη συμβαστική 10. Πέρα τη υποφορία. Εγκρίνεται. 20-16. 361 τώρα. Υπέρ. Α, νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 361. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε προφορίας. 19-17. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 και 362 που είναι ίδιες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 363 Τρασκόφσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 369 Λόκεγάρτ υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά εδώ. 369. Λόκεγάρτ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίες. 19 κατά. Απορρίπτεται συνεπώς. 370. Σάλντο Μόζε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 και 372 που είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 375 έχει αποσυρθεί. 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 379 και 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 383 έχει αποσύρθει. 381 έχει εγκριθεί. 384 είμαστε τώρα στο 384. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 385 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 386 έχει αποσυρθεί. 387 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 388 ως προσθήκη υπέρ υπέρ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 388 ε, 87 88 συγγνώμη ως προσθήκη 388 Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 389 και 390. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67 αποσύρεται. 68 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 391 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 392 αποσύρεται περνάμε στην 393 του κ. Λέκεγκάρτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 καταπίπτει 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 της κυρίας Κόμη και 396 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 397 του κυρίου Λέκεγκαρντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 της κυρίας Κόμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ κατά να το ελέγξουμε να το ελέγξουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι 399 Εγκρίνεται. Η 399 εγκρίνεται. 400. Κυρίου Λέκεγκαρντ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 401 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 402 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 403, συγγνώμη, 401. Να ελέγξουμε την 401, ε, την 402. Ποια θέλετε να ελέγξουμε, την 402, 402. Την είπα λάθος, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 402, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 402 έχει απορριφθεί. Η 401 έχει εγκριθεί. 403. Υπέρ. Υπέρ της 403. Ενδιαφέρον ο συνδυασμός εδώ. Νέος. Ας τη θέσουμε σε ηλεκτρική ψηφοφορία 403. 403. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η 403, 404. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 405. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 73 της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 406 καταπίπτει συνεπώ. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 σχετίζεται με αυτήν. Ψηφίζουμε την 75 λοιπόν. Υπέρ της 75. Κατά. Εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 αποσύρεται. 409 καταπίπτει. 410 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 410 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται συνεπώς. Τροπολογία 77. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά την 411 ελέγχουμε ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία για την 411 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 εναντί 16 17. 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 413 καταπίπτει Συνεπώ. 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 414 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 της συγκήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 416 της κυρίας Στάιλερ υπέρ ανοίγουμε την ψηφοφορία για αυτό της κυρίας Στάιλερ άρχεται η ψηφοφορία για την 4-16 πέρας ψηφοφορίας 12 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται Συμβεστική 13 Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 80 της κυρίας Κόμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 439 του κυρίου Ρέπο υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 81 της κυρίας Κόμη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 442 της κυρίας Χέντ υπέρ κατά να τα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 442 της κυρίας Χέντ πέρας φοφορίας 18 υπέρ 19 κατά καλό είναι που τα ελέγξαμε απορρίπτεται λοιπόν Ψηφίζουμε την 440. 440 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 441 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 443 της κυρίας Χέντ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 444 της κυρίας Χέντ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, ε, εγκρίνεται, συγγνώμη, 82 της κυρίας Κόμη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4.45 του κυρίου Σέλντα και λοιπόν, 4.45 υπέρ, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, την 4.45 νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά, 4.45 του κυρίου Σέλντα και λοιπόν, διάφορες συνδυασμοί, πέρας ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 83 του εισηγήτριας υπέρ, κατά. 446. Παραλείψαμε την 446. 446 ως προσθήκη στην 445. Ως προσθήκη στην 445 υπέρ κατά αποχές δεν είναι καθόλου σαφές. 446. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 17 κατά και μία αποχή. Καλά κάναμε και το ελέγξαμε. 83 της κυρίας Κόμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 της κυρίας Κόμη. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 449 καταπίπτει 447-448 καταπίπτουν 85 της κυρίας Κομή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι λοιπόν καταπίπτουν 452-450 και 451 και φτάνουμε στην 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι λοιπόν καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες. Περνάμε στην 456. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 457 του κ. Σαλβίνη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καθαρά νομίζω. 458 του κ. Σαλβίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 459 του κυρίου Λέκε για κατά αποχές εγκρίνεται 80, 87 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 89 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας ως πρώην ενεργό μέλος. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 90 της κυρίας Κορατσαμπίλτ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 92 του κ. Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά απορρίπτεται 93 του κ. Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 του, της κυρίας Σάλντε Μόσε υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της κυρίας Κόμη απο, έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 2 της κυρίας Κόμη υπέρ κατά εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 της κυρίας Κόμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 της κυρία Κόμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 της κυρία Σαλδεμόσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 του κυρίου Σφάμπα υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ώστε να μην κάνουμε λάθος εγκρίνεται με 19 υπέρ 15 κατά 2 εποχές. Τροπολογία 100 καταπίπτει και η 99 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 107 υπέρ της 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 106 της κυρίας, όχι, λάθος, ε, τροπολογία 6 της κυρίας Κόμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 108 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109 της κυρίας Κορατσαμπίλτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110 της κυρίας Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 111 111 πίπτη, 112 του κύριου Σαλβίνη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Το ελέγξουμε ωστόσο δεν ήταν απολύτως σαφές. Οι φιλελεύθεροι φαίνεται να ψηφίζουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. 112 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, λήξη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 19 κατά. Ε, έπρεπε να το ελέγξουμε λοιπόν. Ένα 13 με κατατμήματα ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ του κυρίου Έγκστρομ. Τμήμα 1 της 113 υπέρ. Κατά αποχές το τμήμα 1 εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Να ελέγξουμε το τμήμα 2 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία το τμήμα 2. Πέρας ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Με 17 υπέρ 19 κατά. 114 του κ. Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 117 του κ. Τσασκόφσκι υπέρ κατά Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 117 του κ. Τρασκόφσκι. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ 16 κατά. Οι 115 λοιπόν και οι 116 καταπίπτουν και ψηφίζουμε τροπολογία 9 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 του κ. Τρασκόφσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 αποσύρεται και 119 θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Την 119 του κυρίου Σουβάμπ και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 του κυρίου Σαλβίνη υπέρ κατά απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 καταπίπτει 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 12 της κυρίας Κόμη υπέρ τροπολογία 12 υπέρ παρακαλώ κατά δεν είναι φες. α εγκρίνεται 128 υπέρ κατά απορρίπτεται Τροπολογία 13 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 13 της κυρίας Κόμη πέρας ψηφοφορίας 18, 18 καλά κάναμε και το ελέγξαμε διότι είναι ισοπαλία απορρίπτεται. Καταπίπτει λοιπόν. Ε, 14 λοιπόν. Υπέρ, κατά. Θα πρέπει να επαναλάβουμε τον έλεγχο για την 14. Τροπολογία 14. Τροπολογία 14. Πέρας ψηφοφορίας 19-18 έχουμε άλλαξε η τακτική εδώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Κάποιο άλλαξε γνώμη μεταξύ τη 13 και 14. 15. Άρχεται η ψηφοφορία για την 15. 18, 19, απορρίπτεται. 13, 14, 15 είναι σαφής. Τώρα 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 του κ. Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της κ. Κόμιος-Προστίκη, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 133 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ειδικά επειδή είναι και δική μου η τροπολογία να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι μεροληπτικός κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 21 υπέρ 15 κατά 134 λοιπόν κατά πίπτη. συμβεστική 3 υπέρ να το ελέγξουμε γιατί δεν είναι όλοι υπέρ. Πάντα είναι καλό να ελέγχουμε τις συμβαστικές υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 19 έναντι 13 και 3 αποχές. 14 κατά, συγγνώμη. Περνάμε στην τροπολογία 19 της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 139 του κ. Σαλβίνη υπέρ κατά εγκρίνεται 20 αποσύρεται, 21 αποσύρεται, 140 της κυρίας Βερνιό υπέρ. Κα, υπέρ, λοιπόν, για την 140 της κυρίας Βερνιό, κατά. Εγ... Να το ελέγξουμε, λοιπόν. 140. 19 υπέρ, 16 κατά. 22 της κυρίας Κόμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 της κυρίας Κόμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογικός 4 της κυρίας Κόμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 141 του κύριου Σφάμπ υπέρ κατά να το ελέγξουμε νομίζω 141 του κυρίου Σφάμπ πέρας ψηφοφορίας 17-16 με τρεις αποχές Μικρή διαφορά. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τελική ψηφοφορία κύριε Σαντεμόζε αποφασίσατε Κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να το σκεφτεί λίγο. Άρχεται η ψηφοφορία για την τελική πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 19 υπέρ, 16 κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολο ήταν αυτός ο φάκελος. Ευχαριστούμε την κυρία Κόμη που μας ε, οδήγησε σε αυτό το σωστό δρόμο, αλλά φυσικά απομένει πολλή δουλειά για να επιτύχουμε μια καλή θέση για το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι έχετε συμβάλει εξαιρετικά σε αυτό. Σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Περνάμε στην επόμενη τελευταία ψηφοφορία που θα είναι πολύ συντομότερη. Πριν από αυτό, ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση, ενώ βρίσκονται όλοι ακόμη εδώ, για να σας πω ότι επρόκειτο να μας επισκεφθεί ο κύριος Κουίν σήμερα το απόγευμα, ο Ιρλανδός Υπουργός αρμόδιος για εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βρίσκεται εδώ στις 3 και ο κύριος Μπρούτον μπορεί να βρίσκεται εδώ στις 3.30 μόνο. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ πριν τις 3.30 ώστε να ξεκινήσουμε ακριβώς τις 3.30 με τον Ιρλανδό Υπουργό. Θα είναι δηλαδή μεγαλύτερο το διάλειμμα σα για το μεσημεριανό, αλλά παρακαλώ να είστε στην ώρα σα και βέβαια βέβαιος ότι θα συμφωνήσει και η κυρία Πρέντεργαστ, γιατί θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε μια όμορφη υποδοχή στου Ιρλανδού συναδέλφου μα σε αυτή την επιτροπή. 3.30 ώρα λοιπόν, αλλά παρακαλώ να είστε εδώ μέχρι τις 3, από τι 3 και 20. Μην τα υπερβολικά. Ας περάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτής τη Επιτροπή ε, προ την Επιτροπή Πολιτισμού για την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Κύριο Γκαρσές Ραμόν είναι ο εισηγητής. δεν είναι εδώ εκ μέρου του. Α, δεν θα μιλήσει κανείς. Σα περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ Νομίζω πως θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Για την τροπολογία 5 είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Όχι, συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Καταπίπτει. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γρήγορα τελειώσαμε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον κύριο Ραμόν και την απουσία του. Πάμε στην οριστική ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Άρχεται η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την επιμονή σας στην ψηφοφορία. Θα σας δώσω στις 3.30 λίγεται η συνεδρίαση.